Good Συνάδελφοι, καλησπέρα. Γίναμε όλο και γυρεότεροι. Είμαι λοιπόν ε, υπεύθυνη για να προεδρεύσω για πρώτη και τελευταία φορά τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Και χαίρομαι που βλέπω φυσιογνωμίες που αναγνωρίζω, να ε, καλωσορίσω και τις καινούργιες φυσιογνωμίες και ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα η επόμενη περίοδος. Ενδιαφέρουσα και γεμάτη πρόκληση. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και θα ακολουθήσουμε το άρθρο 213 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο και στη συνέχεια θα εκλέξουμε τους αντιπροέδρους. Η γραμματεία επίσης ενημερώθηκε για τα αναπληρωματικά μέλη που α, αντικαθιστούν τακτικά μέλη για τη συνεδρία σε αυτή και καταρχάς να υπενθυμίσω ότι έχουμε απαρτία. Ωραία, υπάρχει απαρτία. Υπάρχουν τώρα κάποιοι υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου της ΕΜΚΟ. Ο κύριος Κολάγια. Ε, είναι εδώ. Διερωτώ πως πρέπει να μιλήσουμε τσέχικα. Ο Πέτερ Ντεσούτα είναι ο υποψήφιος που προτείνουμε. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου. Όχι. Η κυρία Ντεσούτερ. Όχι ο κύριος. Κυρία Μπεσούτερ. Έχετε κάποιο πρόβλημα με τον διορισμό? Όχι. Είσαστε πλήρες μέλος, πλήρες μέλος αυτής της Επιτροπής? Ναι. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε ολοκληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και έχετε συμπληρώσει τη δήλωση για τον κώδικα καλής συμπεριφοράς. Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω να διορίσουμε, να ψηφίσουμε μάλλον τον πρόεδρό μας, διαβοής την πρόεδρό μας. Συγχαρητήρια κυρία Ντεσούτερ. Είσαστε η νέα πρόεδρος της Επιτροπής μας. Θα ήθελα λοιπόν να πάρετε αυτή τη θέση. Uh, dear colleagues, thank you very much for Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε για πρόεδρο της Επιτροπής σας. Με μεγάλη χαρά αναλαμβάνω αυτή τη θέση. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά και να προχωρήσουμε τη σημαντική δουλειά αυτή τη Επιτροπή. Είναι καθήκον μου τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, που είναι η εκλογή των αντιπροέδρων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Μας ενημέρωσαν για υποψηφιότητε για διάφορες θέσεις αντιπροέδρων, πρώτο, δεύτερο κτλ. Υπάρχει κάποια αλλαγή στα ονόματα. Λοιπόν, για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου, κυρία Τζενέροβα με μεγάλη χαρά θα προτείνω από το Renew Europe το Pierre Καρλένσκι για την ε, θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και είμαι πεπισμένη ότι θα κάνει θαυμάσια δουλειά. Yes. Μπορώ να ρωτήσω, θα ήθελα να ρωτήσω τον υποψήφιο αν είναι πλήρες μέλος. Ναι, Είμαι, έχετε επίσης ε, συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών ε, συμφερόντων και το κανονισμό για τη δήλωση συμπεριφορά. Ναι. Και συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σας. Ναι. Επομένω, ε, θα ρωτήσω αν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για την θέση του πρώτου αντιπροέδρου και αν δεν υπάρχουν, νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής. Σας καλώ λοιπόν να καθίσετε δίπλα μου στη θέση του Αντιπρόεδρου. Προχωρούμε λοιπόν Κατά τη στοιχεία για τον δεύτερο αντιπρόεδρο υπάρχει υποψηφιότητα. Η κυρία Γκέπχαρτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μεγάλη τιμή εξ ονόματος της ομάδας μου Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να προτείνω την κυρία Μαρία Γκραπίνη. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε. κυρία Γκρατίνη. Ναι, δέχομαι την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα, όλες τις ομάδες. Θα σας ρωτήσω αν είστε πλήρες μέλος της Επιτροπής, αν έχετε συμπληρώσει την δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα και για τη δέσου συμπεριφορά και πόσο το έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη θέση αυτή, όχι. Επομένως, προχωράμε στην ψηφοφορία διαβοής. Προχωρούμε λοιπόν στην θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Αν υπάρχει υποψηφιότητα, ο κύριο Σουάμπ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ουζατούν από την, ε, από την ομάδα EPP. Από ε, ε, το ΕΛΚ, συγγνώμη, δέχεστε την υποψηφιότητα, είστε πλήρες μέλος, ναι, έχετε συμπληρώσει την δήλωση περί οικονομικών συμφερόντων και δέωση της συμπεριφοράς και αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος έχουμε ψηφίσει διαβούλες και έρχεστε στην έδρα. Προχωρούμε τώρα στην θέση του τέταρτου αντιπροέδρου, κύριε Γκέπχαρτ. Κυρία Γκέπχαρτ, ευχαριστώ. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά προτείνω την κυρία Λέιτερ για την υποψηφιότητα αυτή και την δέχομαι. Η κυρία Λέιτα Μάρκετ τη δέχεται την υποψηφιότητα έχετε συμπληρώσει τις ε, αιτήσει ε, που πρέπει για, την οικονομικά συμφέροντα και για δεύσου συμπεριφορά. Ναι. Και τότε διαβοής έχετε τη θέση της τέταρτης αντιπρόεδρου. So now that the uh, Bureau is... Εφόσον λοιπόν ε, έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, ε, σας ανακοινώνω ότι στις 24 Ιουλίου στις 9 το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες θα είναι η, η επόμενη συνεδρίασή μας. Η παρούσα συνεδρίαση λύνεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.